Κυρίε and και κύριοι, καθίστε παρακαλώ και πάλι για να συνεχίσουμε. Έχουμε όχι μόνο την Υποεπιτροπή ασφάλεια και σε αυτό το κομμάτι της συνεδριασιός μας που είναι δημόσια κρόαση, που έχει να κάνει με την κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική και Νότια Συνική θάλασσα και τις επιπτώσεις για την ε, παγκόσμια ασφάλεια. Στην ακρόαση αυτή λοιπόν είμαστε μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την ΑΦΕΤ. Εξού και καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Άντερς Βίστησεν, αντιπρόεδρο της ΑΦΕΤ θα κάνει εκείνο κάποια εισαγωγική παρουσίαση και μετά θα ακούσουμε το πάνελ μας. Έχουμε τέσσερις έμπειρους, εξέχοντες ομιλητές προσκεκλημένους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί όντω έχουμε πολύ σημαντικού ομιλητέ, πιο σημαντικού από μένα. Οπότε σα καλωσορίζω όλου και εκ μέρου τη ΑΦΕΤ και σα ευχαριστούμε πολύ η Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ που μα προσκαλέσατε. Οι εδαφικέ διενέξει στην Ανατολική και Νότια Συνική θάλασσα έχουν να κάνουν ε, όχι μόνο με τις χώρες της περιοχής αλλά και με την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες και σίγουρα μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή και να έχουν επιπτώσει στην ελευθερία ναυσιπλοείας και το εμπόριο. Ανοιχτή σύγκρουση με σημαντικές δυνάμεις μπορεί να έχει απροσδόκητες συνέπειες και είναι και κάτι που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό θα δώσω το λόγο Γιάννα βέβαια στου προσκεκλημένους μας. Εγώ απλώ ήθελα να σας πω πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το θέμα και προσβλέπουμε στη συζήτηση στη συνέχεια. Η κυρία Φωτίνκα. ευχαριστούμε πολύ. Πριν σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας, επιτρέψτε μου στη γλώσσα μου να καλωσορίσω και τους συμπατριώτες μου. Είναι μια πολωνέζικη αντιπροσωπεία εδώ πέρα προσκεκλημένη. Θέλω λοιπόν να σας χαιρετήσω όλους. Πρόκειται για νέους οι οποίοι ήρθαν από την Πολωνία, ήρθαν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, εγώ τους έχω προσκαλέσει. Πρόκειται για νέους διπλωματούχους, δηλαδή πήραν το πολιτήριο φέτος, ε, τελείωσαν το σχολείο και ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτή τη δημόσια ακρόαση όσον αφορά την ασφάλεια στην Ανατολική και Νότια Συνική Θάλασσα. Οπότε και συνεχίζω στα αγγλικά. Λέει η κυρία Φοντίκα, έχουμε τον Γκούναρ Βίγκαντ που είναι ο διαχειριστικός διευθυντής υπεύθυνος για την Ασία και τον Ειρηνικό από την Ευρωπαϊκή Περισσία Εξωτερικής Δράσης, όπως ε, σας τον παρουσίασα και στο προηγούμενο θέμα μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι. Στη συνέχεια έχουμε τον καθηγητή Μπέρναρτ Όξμαν, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. ειδικεύεται στο δίκαιο της θάλασσας. Συνεπώς, η συνεισφορά του στο θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα με τα θέματα νομιμότητας ή όχι στην Ανατολική και Νότια Συνική θάλασσα έχουν μεγάλη σημασία για μας. Στη συνέχεια έχουμε την κυρία Εύα Πέισοβα που είναι αναλύτρια και ερευνήτρια από το Ινστιτούτο Σπουδών Ασφάλειας που δρεύει στο Παρίσι και τέλος έχουμε τον αξιότιμο ερευνητή από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Γκλίγενταλ τον κύριο Φραντς Πολ Φαντερ Πούτεν. Θα συνεισφέρει και αυτός με τη συμμετοχή του στο σημερινό μας θέμα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω λοιπόν το λόγο και θα αρχίσουμε με τον Διευθυντή Βίγκαντ. Παρακαλώ κύριε Βίγκαντ. Mm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να έρθουμε εδώ και να συζητήσουμε μαζί σας αυτό το θέμα που έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια, η περιφερειακή δηλαδή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφής από την αρχή ότι είναι προς το συμφέρον της η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Τέσσερις από τους δέκα βασικούς εταίρους μας είναι στην Ασία, η Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Κορέα. Είναι τεράστιες ε, οι ποσότητες εμπορευμάτων που περνούν από την θάλασσα αυτή. Γι' αυτό και αυτή η θάλασσα έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλες τις οικονομίες και για εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα που για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να ε, κατασκευάσει διάφορα προϊόντα που κατασκευάζει, μην έχοντας ε, τις προμήθειες οι οποίες περνάνε από τη θάλασσα αυτή, αν τυχόν είχε κλείσει αυτή η θάλασσα. Συνεπώς, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει. Και θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Η παγκόσμια στρατηγική λοιπόν που ενέκρινε το Συμβούλιο το 2016, τον Οκτώβριο, λέει σαφώ ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ασία αποτελούν προπόθεση για την ευημερία μας. Είναι προ το συμφέρον μας να ενισχύσουμε τις διπλωματικέ μας σχέσεις με την Ασία. Τώρα πιο συγκεκριμένα για την Ανατολική και Νότια Συνική θάλασσα, θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε μία δήλωση που έκανε το Μάρτιο, είπα, εκπρόσωπος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι σημαίνει δήλωση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ των 28 χωρών μελών. Και λέει το εξή. Ρητά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανησυχεί για την εξάπλωση των πυράβλων στην ε, νότια και ανατολική συνική θάλασσα. Ο επέκταση του εξοπλισμού αυτού μπορεί να απειλήσει την ελευθερία αναυσιπλοείας ή τις ελεύθερες πτήσεις, κάτι το οποίο μας ανασυχεί όλους ιδιαίτερως. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από όλες τις ελευθερες πτησεις κατι το οποιο μα ανασυχει ολου ιδιαιτερως συνεπως η ευρωπαικη ενωση ζητα απο ολες τις πλευρες που έχουν διεκδικήσει να επιδείξουν συγκράτηση και να μην προχωρήσουν σε μονομερείς δράσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ των 28 ε, μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου τον Ιούλιο. Βέβαια, τα θέματα αυτά μας απασχολούν ήδη από πολύ πριν. Το 2012, για παράδειγμα, υπήρξαν κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την διένεξη στη θάλασσα αυτή. Και δυστυχώς η κατάσταση παραμένει ίδια μέχρι σήμερα. Έχουμε και την στρατηγική μας για την Κίνα, τη στρατηγική μας για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά από την διάσκεψη με την Κίνα και την απόφαση του δικαστηρίου και δύο δηλώσεις, τη μία από τις οποίες σας τη διάβασα. Οι βασικές αρχές αναφέρονται σε αυτές ακριβώς τις θέσεις. Πρώτον, όσον αφορά την σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται για τη διατήρηση του δίκαιου της θάλασσας βάσει της αρχής του διεθνούς δικαίου, βάσει της σύμβασης και της αρχής της ειρηνικής πύλησης διανέξεων. Όσον αφορά τώρα την Ανατολική και Νότια Συνική Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτήν, γιατί θέλει να προωθήσει τις αρχές που αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο, την ελευθερία ναυσιπλοείας και την μείωση των εντάσεων που μπορεί να επηρεάσουν τις επενδύσεις στο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και όχι μόνο. Τρίτον, για διεκδικήσεις και επίλυση διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τοποθετείται όσον αφορά τα θέματα κυριαρχία που έχουν να κάνουν με εδαφικέ διεκδικήσεις. Συγχρόνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να λύσουν τις διαφορές τους και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με ειρηνικό τρόπο και με συνεργασία. Και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο συμπεριλαμβάνει τη Σύμβαση για το Δίκαιο στη Θάλασσα, την UN Clause και τις διαδικασίες διαιτησίες βέβαια στα πλαίσια αυτής. Στηρίζει τις περιφερειακές διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει την κατάληξη των συνομιλιών για ένα κώδικα διοντολογίας μεταξύ των χωρών ΑΣΕΑΝ και της Κίνες μετά την δήλωση του 2002 για την διαδολογία των μερών στην περιοχή. Ο κώδικας διοντολογίας θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την στήριξη Τη περιφερειακή και διεθνούς τάξη. Τώρα, προκειμένου όλε αυτές τι αρχές να υλοποιηθούν, να γίνουν δράση, έχουν αναλυφθεί οι εξή πρωτοβουλίε μέχρι τώρα. Τον Νοέμβριο του 2013 ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει τον πρώτο διάλογο υψηλού επίπεδου σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, διέλευση στην θάλασσα. Είχε να κάνει με την ε, επίβλεψη στη θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να προσφέρει στους εταίρους ΑΣΕΑΝ όσον αφορά την κοινή διαχείριση των πόρων. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και μεταξύ των χωρών μελών μας. Ό,τι διαφορές υπάρχουν ε, μεταξύ των χωρών μας δεν έχουν όλες επιληθεί, αλλά πολλές ναι, μεταξύ ε, κατοχωρών και Γερμανίας για παράδειγμα. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Βιετνάμ για την Αυστραλία θα αναλάβουν την Προεδρία της περιφερειακής ΑΣΕΑΝ όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας για τα επόμενα τρία χρόνια από το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Προετοιμάζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας που έχει να κάνει με την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, το περιβάλλον, την ανάπτυξη αλλά και τη συνεργασία βάσει του κράτους δικαίου. Τέλο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί από κοντά τη νομοθετική διαδικασία σε χώρες εταίρου στην Ασία που επηρεάζουν ε, τα θέματα της ναυσιπλοεία και τη δικαιοδοσία στην ναυσιπλοεία. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας τώρα στον νόμο της Κίνας για την ανοιχτή θάλασσα. Μαζί με χώρες όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε κάνει σχόλια για τις τροπολογίες στην νομοθεσία αυτή του 84 και λέμε ότι η νομοθεσία πρέπει να παραμείνει να συμμορφώνεται με τις αρχές της UN CLOS, δηλαδή της Σύμβασης για το Δίκαιο στη Θάλασσα. Έχουμε όπου να είναι και την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, αρχές Ιουνίου. Επί τη ευκαιρία αυτή θα ανακηρύξουμε το έτος των επαφών μας με την Κίνα όσον αφορά τη θάλασσα και θα επικεντρωθούμε σε θέματα διακυβέρνηση των ωκεανών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίγκαν, κύριε Φιντά. Καθηγητά Όξμαν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε κυρία Προέδρη, δικαιοκριμένο αντιπρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, δικαιοκριμένα μέλη. Μεγάλη τιμή για μένα που προσεκλήθη να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Το κάνω αυτό υπό την ιδιότητά μου που εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό προσωπικά. Μιλώντας σε μια δεξίωση για τον απερχόμενο νομικό σύμβουλο, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών Χένικ Κίσιγκερ εκμυστηρεύτηκε ότι αυτό που εκτιμούσε περισσότερο σε ένα νομικό ήταν ότι ε, του υπενθύμιζε τη βάση της αρχές από την οποία στεκόμαστε. Ειδικά όταν ε, δεν ήθελε να το ακούσει αυτό. Η πλατφόρμα της αρχής που θα πρέπει να διέπει την προσέγγιση μας στα προβλήματα τα οποία συζητούμε στην ακρόαση είναι το κράτος δικαίου ε, στα διεθνή ζητήματα όπως μας τόνισε μόλις τώρα και ο Σβίγκαν, αυτό αποτελεί και θα πρέπει να αποτελεί ε, το δώρο, το βιώσιμο τη διαρκείας ε, της Ευρώπης ε, για την Ευρώπη και τον κόσμο στη γη και στη θάλασσα. Οι του πυλώνες του σύγχρονου, της συγχρόνου ενόμου τάξης ωκεανούς είναι η χάρτα του ΟΗΕ και η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αμέλεια και παράβαση ουδήποτε από αυτά τα δύο νομικά κείμενα ίσως να εκδηλωθεί σαν ένα περιφερειακό πρόβλημα με συνέπειες για την όλη περιοχή. Αλλά οι παγκόσμιες συνέπειες τέτοιας ασέβειας για αυτή την νομοθεσία θα πρέπει να είναι σαφής. Δηλαδή αποτέλεσμα είναι η αποδυνάμωση της διεθνούς ενόμου τάξους, συνεπώς και μια αποδυνάμωση της ε, παγκόσμιας ασφάλειας. Οι αξιώσεις και οι διεκδικήσεις της Κίνας στη νότια συνική θάλασσα και οι δράσεις που απορρέουν από αυτό ε, αποτελούν μια πρόκληση σχετικά με αυτό. Ισχυρίζεται ότι η Κίνα, ότι τα θέματα που τίθενται είναι περιφερειακά και θα πρέπει να επιληθούν από τις χώρες της περιοχής. Αυτό πράγματι ισχύει. Αλλά οι διεκδικήσεις της Κίνας και οι σχετικές δράσεις εν τη επιδιώξη των στόχων ε, εμπλέκουν δύο συμφέροντα όλων των κρατών είτε έχουν σύνορα είτε δεν έχουν σύνορα με την Νότια Συνική Θάλασσα. Καταρχάς αφορά το συμφέρον για τη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας και ειρήνης και της ειρηνικής διευθέτησης των διεθνών διαφορών σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτό το συμφέρον είναι στο επίκεντρο του στόχου και του σκοπού της Χάρτας του, των Ηνωμένων Εθνών. Δεύτερον, είναι το συμφέρον να εξασφαλίζουμε παγκόσμια τάξη στι θάλασσε και του ωκεανού. Αυτό συμπεριλαμβάνει το σεβασμό των εταιριών και δικαιωμάτων τη ναυσιπλοεία και τη επικοινωνία που απολαμβάνουν όλε οι χώρε, καθώ και το καθήκον για την προστασία και τη διατήρηση του θαλασσιού περιβάλλοντο. Και αυτό σε όλα τα μέρη, σε όλε τι θάλασσε. Αυτό το συμφέρον είναι στο επίκεντρο του στόχου και του σκοπού τη συμβάσεω του ΙΕ για το δίκαιο των θαλασσών οι προκλήσει και τα προβλήματα για οποιοδήποτε αυτά τα συμφέροντα πιθανότατα η μία πτυχή είναι επηρεάζει την άλλη. Η παγκόσμια κινητικότητα στις θάλασσε είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας και σταθερότητας. Δοθήσεις της επιλογής, καμία χώρα δεν θα ανεχθεί παρέμβαση ε, όσον αφορά τι ζωτικέ γραμμέ επικοινωνία που διαθέτει αυτή η χώρα. Οι προκλήσει σε οποιοδήποτε συμφέρον αυτό σε κάποιο τμήμα του κόσμου, αν δεν ελεγχθεί και δεν επιληθεί, δημιουργεί και άλλες προκλήσεις σε αυτά τα συμφέροντα σε άλλα σημεία της υδρογείου. Να σας παρουσιάσω αυτό το θέμα συγκεκριμένα με τις διεκδικήσεις που έχει η Κίνα. Καταρχάς η Κίνα διεκδικεί ιστορικά δικαιώματα σε τεράστιο τμήμα της νότιας συνικής θάλασσας. Αυτή η διεκδίκηση συνδέεται με την όπως αποκαλούμενη ε, γραμμή, με γραμμές που έχει χαράξει η Κίνα. Βλέπετε τις διακεκομένες γραμμές ε, με κόκκινο στο χάρτη στην οθόνη σας. Λοιπόν, διεκδικεί ιστορικά δικαιώματα η Κίνα, αλλά αυτό δεν βασίζεται στα δικαιώματα που απορρέουν από τη Σύμβαση για το Δίκαιο των Θαλασσών και θέλει να παρεκκλήσει από τα δικαιώματα άλλων χωρών δυνάμει της συμβάσεως αυτής. Η απόφαση λοιπόν για, του Διευθυντικού Δικαστηρίου για την Νότια Συνική Θάλασσα συμπεραίνει ότι υπερισχύει ο νόμος ε, της συμβάσεως για τις θάλασσες προτέρων διεκδικήσεων και ε, ε, εν πάση περιπτώσει και οι άλλες ε, ενδιαφερόμενες χώρες δεν συμφώνησαν με τις διεκδικήσεις της Κίνας βάσει ιστορικών δικαιωμάτων. Όμως ρητά η Κίνα επανειλημμένα έχει διεκδικήσει ιστορικά δικαιώματα που έχει στην νότια Συνική θάλασσα μετά την απόφαση που απέρριπτε τους ισχυρισμούς της. Αυτό δημιουργεί μια πρόκληση και πρόβλημα όσον αφορά τη διεθνή ενόμη τάξη. Οι χώρες που προηγουμένως ε, προέβαλαν διεκδικησει που ξεπέρναγαν τα όρια που προβλέπει η Σύμβαση για το Δίκαιο των Θαλασσών, προέβαλαν, ε, μάλλον συμμόρφωσαν τι διεκδικήσει του με την Σύμβαση από όταν έγιναν συμβαλόμενα μέρη. Η Κίνα έκανε ακριβώ το αντίθετο. Και αν η Κίνα μπορεί να το κάνει αυτό και άλλοι ίσως να ακολουθήσουν. Πολλέ χώρε, πολλές χώρες έχουν μακρά ιστορία ε, επαφής ε, με τη θάλασσα, χρήση της θάλασσας και διεκδικήσεις όσον αφορά τις θαλάσσιες Βεβαίως ε, και πολύ λογικά κάποιες χώρες αραβικών χωρών αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τον όρο περσικός κόλπος. Ακόμα κι αν ε, δεχτούμε τις διαβεβαιώσει τη Κίνας ότι οι ιστορικές της διεκδικήσεις δεν έχουν πρόθεση να επηρεάσουν την ελευθερία της ναυσιπλοεία, η αποδυνάμωση της ενώμη τάξη που δημιουργείται από τη Σύμβαση σαν αποκλειστική βάση για αξιώσει όσον αφορά τι θάλασσε αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων όσον αφορά την ελευθερία ε, ναυσιπλοείας αλλού στον κόσμο. Δεν θα ήταν δύσκολο να βρει κανεί νομικού που φρονούν ότι η ελευθερία τη ναυσιπλοεία επηρεάζεται από ιστορική φύσεω διεκδικήσει, ιστορικέ διεκδικήσει. Πέρα από αυτή την αξίωση βάσει ιστορικών ε, δικαιωμάτων, η Κίνα ισχυρίζεται ότι οι νήσοι Σπράτλι παράγουν ε, μία σειρά δικαιωμάτων στη θάλασσα όταν, όπως πιστεύει η Κίνα, εξεταστούν ως ένα σύνολο. Αυτή η θέση απερίφθη ε, στην απόφαση τη δυτική για την Νότια Συνική Θάλασσα, αλλά τώρα προβάλλεται όλο και περισσότερο από κινέζικες πηγές μετά τη ληφθήσα αυτή η απόφαση. Αυτό δεν είναι απλώς, και το τονίζω, απλώς τεχνικό ζήτημα ε, νόμου των θαλασσών. Η σύμβαση επιτρέπει μόνο χώρες με αρχιπέλαγος που απαρτίζονται αποκλειστικά από νήσους κράτη αρχιπέλαγα να χαράξουν ε, ε, γραμμές που περικλείουν τα ύδατα μιας υπεράκτιας νησιωτικής ομάδας και να θεωρηθεί αυτός ο αρχιπέλαγος. Επιβάλλεται αυτή η αρχή από τη σύμβαση λόγω της ανησυχίας ότι αν οι πυρωτικές χώρες επιτρεπόταν να περικλείσουν τα ύδατα ε, με εντός υπερακτίων ισιωτικών ομάδων και θεωρηθούν αυτά εσωτερικά ύδατα, αυτό θα υπονόμευε την ελευθερία της ε, και των υπεπτήσεων και συνεπώς θα μπορούσε αυτό να απειλήσει τη διεθνή ειρήνη ε, και την ασφάλεια. Δεν χρειάζεται κανείς να κοιτάξει μακριά, ας δείξουμε ματιά στο Αιγαίο για να εκτιμήσει και να καταλάβει αυτές τις ανησυχίες. Λοιπόν, η βάση των αξιώσεων σύμφωνα τις οποίες οι νήσοι Σπράτλι μπορεί να περικλειστούν και να θεωρηθούν σαν ομάδα, σαν συστάδα νησιών, ε, είναι εθιμικό διεθνές δίκαιο. Αυτή η λογική, αυτή καθεαυτή, δημιουργεί συστημικό κινδυνό, απειλή όσον αφορά τη σύμβαση του νόμου των θαλασσών και απειλή και τις πολ, ε, πολυμερείς παγκόσμιες συμφωνίες σαν αποκριστική βάση ε, για ε, καθορισμό κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θάλασσα. Ο σκοπός της συμβάσεως για το δίκαιο των θαλασσών ήταν να ξεπεραστεί η αστάθεια και η αβεβαιότητα που αναπτύχθηκε όταν μονομερείς αξιώσεις ε, για θάλασσες ε, πολλαπλασιάστηκαν τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αν δεχτούμε την έννοια σύμφωνα την οποία αυτή η διαδικασία μπορεί τώρα να συνεχιστεί εν παρεκκλήση της συμβάσεως και των διατάξεων αυτής, είναι απίθανο ότι αυτός ο κατακαιρματισμός και τα προβλήματα θα περιοριστούν σε συστάδες ε, νησιωτικές. Μία από τις πιο σημαντικές συνεισφορές της συμβάσεως των θαλασσών στο κράτος δικαίου σε διεθνείς σχέσεις είναι η συμπερίληψη διατάξεων που δίνει σε οποιοδήποτε μέρος που έχει διαφορές όσον αφορά τη σύμβαση στο δικαίωμα να ε, καταφύγει σε διαιτητική λύση, σε διαιτησία. Όλα τα μέρη της συμβάσεως έχουν συμφωνήσει ε, γίνοντας μέλη της συμβάσεως. Εάν αν είμαστε σοβαροί για το κάτω δικαίου όσον αφορά τι διεθνεί υποθέσει, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί όσον αφορά το καθήκον να σεβόμαστε νομικά δεσμεύουσε δεσμεύουσες αποφάσεις. Όμως η Κίνα ρητά απορρίπτει, απορρίπτει συγγνώμη, αυτή την απόφαση, προβάλλει ισχυρισμού που απερίφθησαν κατά τη διαιτησία και αντίθετα από άλλε χώρε σε ανάλογε περιστάσει μέχρι τώρα δεν δείχνει σαφή σημάδια ότι στην πράξη ε, συμμορφώνεται. Πρέπει να είμαστε επίσης σαφείς για τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ δικαιώματος από τη μία πλευρά και αμφισβητούμενες ε, επικράτειες αμφισβητουμένων ορίων μεταξύ χωρών από την άλλη. Τα τελευταία αυτά θέματα μπορούν να ε, λυθούν από τις χώρες που έχουν τέτοια προβλήματα ε, και ε, ε, ίσως να είναι θέματα που άλλα κράτη δεν δέχονται να τοποθετηθούν από αυτόν, όπως είπε και ο Σβίγκαν. Αλλά Το θέμα ότι κατά πόσο έχει δικαίωμα μια χώρα να διεκδικήσει κυριαρχία, κυρίαρχα δικαιώματα για ένα τμήμα της θαλάσσης ή της υφαλοκρηπίδας ή του βυθού και αν, σε ποιο βαθμό και πού, είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις χώρες. Επηρεάζει τα δικαιώματα που έχουν, τις ελευθερίες τους και τα συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας στο σύνολό της. Έτσι, επί παραδείγματι, η Κίνα δημοσία έχει αμφισβητήσει τα δικαιώματα της Ιαπωνίας σε αδίποτε δικαιώματα υφαλοκρηπίδας όσον αφορά ε, το ο κύριο Τόμ Σίμα θεωρώντας ότι είναι απλώς ε, βράχος, βραχονισίδα και αυτό το θέμα είναι κάτι που προβληματίζει τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Στη Νότια Συνική Θάλασσα, στη Διαιτησία, ε, το δικαστήριο αντιμετώπισε παρόμοιο θέμα. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε από, από τα νησιά του Σπράτλι έχουν δικαίωμα αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαροκρηπίδα, ε, πέρα από τα ε, χωρικά ύδατα. Αποφασίστηκε από τη δική αρχή ότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μικρά τα νησιά αυτά τα Σπράτλι. Το μεγαλύτερο είναι μικρότερο από μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αν όλα τα πάρουμε μαζί, θα ήταν σαν τον Μπουάντε Μπουλόνι στο Παρίσι. Αλλά η παρουσία μικρών χαρακτηριστικών τέτοιων σε ημιπεριήκλειστες θαλάσσιες περιοχές μπορεί να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τις ε, γειτονικές χώρες. Ας σας δείξω κάποια διαγράμματα για να καταλάβετε. Στην οθόνη βλέπετε ε, μία εκπροσώπηση τριών χωρών που ε, είναι γύρω από μία ημίκλειστη θαλάσσια περιοχή. Προσθέτουμε τώρα 12 ε, μίλια χωρικά ύδατα ε, για κάθε μια τέτοια οντότητα. Προσθέτουμε και 200 μίλια αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα ε, για κάθε μία από αυτές τις χώρες. Υποτεθείστε τώρα ότι υπάρχει ένα μικρό νησάκι στη μέση που τελεί υπό την κυριαρχία άλλης χώρας. Αυτό το νησί παράγει χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων. Τώρα θα υποθέσουμε ε, τρία πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ότι αυτό το νησάκι, το πολύ μικρό νησάκι, ενδεχομένως, και το λέω αυτό υποθετικά, ε, θεωρείται ότι είναι ένα πλήρες δικαιούχο νησί και όχι βραχό νησίδα. Άρα είχε δικαίωμα να έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα ε, σε ακτίνα 200 ναυτικών μιλίων. Δεύτερον, ότι δεν υπήρχε σαφής οριοθέτηση επικάλυψης ε, δικαιωμάτων στη ζώνη αυτή των 200 μιλίων. Και τρίτον, ότι αυτή η χώρα που έχει την κυριαρχία πάνω σε αυτό το μικρό νησάκι θα διεκδικήσει και θα εφαρμόσει τα αποκλειστικά κυρίαρχα δικαιώματα και δικαιοδοσία σε όλες τις ζώνες των 200 μιλίων που γεννώνται από αυτό το μικρό νησάκι χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα άλλων χωρών, των άλλων γειτονικών χωρών. Ιδού το αποτέλεσμα. θα πρέπει όλοι να θαρρυνθούμε από αναφορές ότι επιτυγχάνεται πρόοδος από την Κίνα και τις χώρες ΑΖΕΑΝ συντάσσοντας, ετοιμάζοντας ένα πλαίσιο για ενδεχόμενο διοντολογικό κώδικα που θα είναι νομικά δεσμευτικός. Πρέπει επίσης όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν απαλλάσσει την Κίνα από τα νομικά καθήκοντα που υπέχει από την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και τον νόμο των θαλασσών και σχετική σύμβαση. Άρα έχει μεγαλύτερο κίνητρο πιθανόν η Κίνα να συνάψει και να εφαρμόσει ε, έναν ε, διοντολογικό κώδικα που έχει νόημα και να βοηθήσει τις αρχές της να αντισταθούν σε πιέσεις εκείνους που θέλουν μια πιο αδιάλακτη συμπεριφορά. Το να γίνει σαφές το μήνυμα μας κάνει να αποφύγουμε τον κίνδυνο ότι η σιωπή θεωρείται από την Κίνα ή από οποιοδήποτε άλλον σαν συμφωνία, σαν συνένεση. Θα μπορούσα να προσθέσω ότι αυτό το μήνυμα είναι προς όφελος μακροπρόθεσμο της ε, Κίνας. Η Κίνα είναι μια αναδυόμενη θαλάσσια δύναμη. Την συμφέρει σταθερότητα όσον αφορά τον νόμο των θαλασσών Τη συμφέρουν οι παγκόσμιε ελευθερίε τη ναυσιπλοεία και των επικοινωνιών και τα συμφέροντά τη αυτή θα αυξάνουν την πρόοδο του χρόνου. Αυτό το αυξανόμενο συμφέρον, δηλαδή να εξασφαλίζει ε, τα νομικά δικαιώματα και υποχρεώσει όλων των κρατών μελών σύμφωνα τη Σύμβαση του Δικαιώματο των Δασών, θα ενισχύεται από τι προσδοκίε συμμόρφωση μεταξύ των πιο σημαντικών διεθνών παικτών. Άρα έτσι θα είναι πιο εύκολο για την Κίνα, όπως και άλλες χώρες πριν από αυτήν, να βρει και τη βούληση να προσπαθήσει να υπερκεράσει τις, τις παραβάσεις που κάνει. Λοιπόν, συμπεραίνω ότι οι προπτικές για την αποφυγή της αποδύναμης του διεθνούς νόμου και στην Νότια Συνική Θάλασσα και αλλού θα βοηθηθεί και θα διευρυνθεί από σαφείς ενδείξεις ότι η Κίνα αναμένεται να συμμορφωθεί με τις διεθνείς υποχρεώσεις δυνάμει της Χάτας των Εθνών και της Συμβάσεως για τον νόμο των θαλασσών και ότι αυτό συμπεριλαμβάνει δύο πράγματα όλος ιδιαίτερος. Ήτι περιορισμό των θαλασσίων διεκδικήσεών της στα δικαιώματα που έχει και που απορρέουν από τη σύμβαση του νόμου των θαλασσών και ότι θα σέβεται τα δικαιώματα και ελευθερίες, ναυσιπλοή και τα άλλα δικαιώματα όλων των χωρών δυνάμει της συμβάσεως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Και τώρα δίνω το λόγο στη δόκτωρα Εύα Πέχσοβα από το EUISS. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Έκλεισε το μικρόφωνο. Ε, μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις συνέπειες των εντάσεων στην ασφάλεια και αυτή είναι η πρόθεσή μου. Θα δω συγκεκριμένα τις στρατηγικές επιπτώσεις των εξελίξεων σήμερα, γεωπολιτικό αντίχτυπο των εντάσεων, και τα οικονομικά συμφέροντα. Σκόπιμα άφησα τις πολύ σημαντικές νομικές επιπτώσεις αφού ήξερα ότι ο καθηγητής Όξμαν θα τις εκάλυπτε αυτές. Ε, τα πιο σημαντικά θέματα τα ανέφερε. Καταρχήν ένας χάρτης χρειάζεται, παρόλο που γνωρίζετε τα βασικά προβλήματα στην Ανατολική και Νότια Κινέζικη θάλασσα τονίζω ότι εκτός από το 90% ε, της διεκδικήσεις της ε, Κίνας, 11 και 9 παύλες, ε, υπάρχουν και άλλες διεκδικήσεις από την Ιαπωνία, την, τις Φιλιππίνες, αλλά και πιο μικρές Μπρουνέι, από Μπρουνέι κλπ. Επίσης, οι διαφορές δεν είναι καινούριε ε, από, από μνημόνευτα χρόνια, α, όχι από μνημόνευτα, αλλά πολύ παλιά πάντως υπάρχουν διαφορές εδώ. Τώρα τελευταία προσέξαμε περισσότερο το θέμα μετά το 2009, δηλαδή ε, όταν κινήθηκε νομικά η Κίνα. Γιατί για πρώτη φορά τότε επίσημα αναδεικνύεται η γραμμή των 9 παυλών ως επίσημο κινέζικο αίτημα. Και μετά το 2013 ε, όταν ε, ε, προσέφηκαν και οι Φιλιππίνες στο Διεθνές Δικαστήριο, έχουμε αποδείξεις ότι σχηματίζει, κατασκευάζει νησιά η Κίνα στα Σπράτλι που είναι τα πλέον διαφιλονικούμενα. Όπως είπε ο καθηγητής Όξμαν, πέρσι υπήρξε απόφαση και τώρα μπορούμε να προβάλλουμε την απόφαση αυτή χωρίς να σημαίνει ότι η διαφορά εξαφανίζεται. Ε, εδώ βλέπουμε δορυφορικές ε, λήψεις ε, από το Νοέμβριο 2016, από το 2013 και πριν, λίγο πριν, άρχισε η Κίνα ε, να ε, δημιουργεί εδάφη ε, με, δημιουργώντας, δημιουργώντας νησιά ή μεγαλώνοντάς τα βλέπουμε εδώ διάφορους, διάφορες βραχονησίδες το πιο σημαντικό στις εικόνες αυτές είναι η στρατιωτική σημασία των εγκαταστάσεων που φαίνονται εκεί και συγκεκριμένα ε, ε, τα σημεία προσγείωσης, ε, οι διάδρομοι προσγείωσης, υπάρχουν μεγάλες αποθήκες, χάγκαρ και έχουμε και συστήματα πυραυλικά, εδάφους, αέρος που δημιουργούν υποψίες σε σχέση με τις προθέσεις της Κίνας. Συχνά αναφέρεται ότι η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα που δημιουργεί νησιά. Αλήθεια είναι αυτό. Ε, αλλά για να έχουμε κάποια αίσθηση του μέτρου, εδώ έχουμε προσπάθειες από το Βιετνάμ για κα, κάτι τέτοιο σε πολύ μικρότερο βαθμό ε, διάδρομο προσγείωση έχει ένα νησί. Και για να δείτε εδώ τις συγκρίσεις ε, τα τελευταία χρόνια, η, η Κίνα ε, πήρε, προσέθεσε 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ το Βιετνάμ 120 μόνο. Η ο, διάδρομ, ο διάδρομος προσγείωσης και το μήκος του μας δείχνει και τι ε, ε, ε, αεροπλάνα μπορούν να εξυπηρετηθούν εκεί. Δεξιά, στο Fury Cross, υπάρχει ένας διάδρομος προσγείωσης που μπορεί να εξυπηρετήσει βομβαρδιστικά και αυτό οπωσδήποτε κάνει μια ειδοποιό διαφορά. Τώρα, τα σπράτλη τώρα. Η κίτρινες κουκίδες, οι 7 είναι νησιά της Κίνας, τα κόκκινα είναι του Βιετνάμ, ορισμένα είναι μαλαισιανά, αλλά αυτά δεν είναι καινούρια. Αυτό που συμβαίνει πρόσφατα και μέχρι και την περασμένη Παρασκευή ήταν η ανακοίνωση της Κίνας της πρόθεσής της να ε, κάνει κατασκευές και στα, στη βραχονισίδα Σκάρμπορο. Αυτό οι αναλυτές το παρακολουθούν και προειδοποιούν ε, έναντι του κινδύνου αυτού εδώ και χρόνια. Έχει σημασία η βραχονισίδα Σκάρμπορο, στρατηγική σημασία, όπως βλέπετε και στο χάρτη ήταν ε, το, η τελευταία κίνηση που θα έκανε η Κίνα για να έχει πλήρη έλεγχο της νότιας κινέζικης θάλασσας ε, που θα της επιτρέψει να καλύψει ε, και ένα αέριο χώρο. Αυτό δεν το λέω για να φοβήσω, αλλά για να παρουσιάσω κάποια στοιχεία. Σε περίπτωση που κάποιος θα σκεφτόταν ότι... Δηλαδή, εάν προτίθετο η Κίνα να ε, ανακηρύξει μία ζώνη ε, αμυντική ε, στην περιοχή αυτή, η ε, βραχονισίδα Σκάρμπορο το επιτρέπει να το κάνει. Μέχρι τώρα είχε περιβαλλοντικό σταθμό παρακολούθησης στο Σκάρμπορο. Συνήθως έτσι άρχιζε η Κίνα. Το... Όταν άρχισε να δημιουργείται το Fury Cross, το ίδιο πρόσχημα προευλήθη και βλέπετε τι συνέχεια δόθηκε και τι μορφή έχει σήμερα. Τώρα, η δραστηριότητα της Κίνας στην Νότια Κινέζικη θάλασσα. Έχει απασχολήσει και πέρσι το Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχουν ε, σαφείς απειλές. Μπορούμε να δούμε ε, κάποιους ε, ορισμούς για τον υβριδικό κίνδυνο. Ε, βλέπουμε ότι ε, υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Υπάρχουν μη συμβατικές μέθοδοι. Η Κίνα χρησιμοποιεί μη στρατιωτικές μεθόδους, ε, χρησιμοποιεί την ακτοφυλακή της, τον αλλιευτικό στόλο της, ε, που τυχαίνει να είναι οπλισμένος. Ε, επίσης χρησιμοποιεί, κάνει πολύ έξυπνα μικρά βήματα, σαλαμοποίησης που είναι, ε, έτσι το, τα λέμε, είναι δύσκολο να τα δούμε. Η, συμπεριλαμβάνεται η, η νότια κινέζικη θάλασσα σε μια ευρύτερη ε, διοίκηση ε, που διαχειρίζεται όλη αυτή τη τεράστια περιοχή. Επίσης έχουμε ανάπτυξη του τουρισμού, ε, κρουαζιερόπλια. Δημιουργείται δηλαδή τετελεσμένο γεγονός στην νότια Κινέζικη θάλασσα που δύσκολα θα ανατραπεί. Η ε, Κίνα πάντοτε προτιμούσε διμερείς διαπραγματεύσεις με τις χώρες που είχαν διεκδικήσει στις Φιλιππίνες, στο Βιετνάμ και πάντα ε, χρησιμοποιεί ε, διπλωματικούς τρόπους συζητήσεων αλλά και εμπορικά κίνητρα. Βέβαια η λέξη bullying, εκφοβισμός, θα ήταν πολύ ε, βαριά λέξη εν προκειμένου. Ε, τώρα, για το, υπάρχει κεντρικός συντονισμός, στην Κίνα αυτό είναι σαφές, οι στόχοι είναι σαφείς ε, θέλει να επιβληθεί το Πεκίνο εκεί. Είναι ε, θέμα εθνικών συμφερόντων ετώ. Αυτό διαπραγματεύεται και δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών στη νότια κινέζικη θάλασσα όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Ε, το τελευταίο είναι το πιο ανησυχητικό. Είναι δηλαδή αυτή η αμφισημία ε, στις, στους ισχυρισμούς της Κίνας. Ε, Επίση, η απόκτηση των, της βραχονισίδας είναι ένα άλλο στοιχείο. Το 2016 ε, όταν έγιναν προσπάθειες ε, μεταξύ, μεταξύ Φιλιππίνων και Κίνας, το Σκάρμπορο ήταν μια βραχονισίδα που δεν έπρεπε να συζητηθεί. Και ένα χρόνο αργότερα ε, βλέπουμε τη σημερινή κατάσταση, πώς διαμορφώθηκε αυτό, δημιουργεί απογοήτευση και μας κάνει να μην ε, μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά της Κίνας. Βέβαια, οι εντάσεις στην Νότια Κινέζικη θάλασσα ε, αύξησαν σημαντικά τις πιέσεις ε, στη δυναμική σε περιφερειακό επίπεδο για την ασφάλεια. Ε, οι ΙΠΑ ε, έχουν παλιά στρατιωτική παρουσία, ε, έχουν ελευθερία αναυσιπλοείας για τις επιχειρήσεις τους, αλλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πολλοί αμφισβητούν την νομιμοποίηση της παρουσίας των ΗΠΑ δεδομένων των εξελίξεων σήμερα που δεν μπόρεσαν να ανασχεθούν από τη ΣΥΠΑ. Η Ιαπωνία έχει ζωτικά συμφέροντα στην Νότια Κινέζικη θάλασσα και ήταν από τα μέρη που άρθρωσαν ε, χειρό λόγο ε, ε επίσης ε, αύξησαν την στρατιωτική τους παρουσία και τα σύγχρονα σκάφη στην Νότια Κινέζικη θάλασσα για να συνενωθούν ε, και να κάνουν, και να κάνουν κοινές ασκήσεις ε, με ε, Ινδονησία και είπα. αυτά η Κίνα τα παρακολουθεί εκ του σύνεγγης. παρακολουθώντας το ενδεχόμενο διεθνοποίησης του θέματος που θα επηρέαζε ενδεχομένως τις δικές τους διεκδικήσεις. Η ΑΣΕΑΝ πλήττεται ε, πολύ περισσότερο πέρα από τις διμερείς επαφές η Κίνα πάει να διαλύσει την ΑΣΕΑΝ εδώ αποδυναμώνεται η αρχιτεκτονική της περιοχής γιατί η ΑΣΕΑΝ ε, είναι ένας φορέας που μπορεί να παίξει ρόλο για την ε, ασφάλεια και έχουμε και την Ινδία τους άλλους χρήστες η Ινδία ενέχεται περισσότερο. Η Αυστραλία έστειλε πλοία επίσης στην Νοτιοκινέζικη θάλασσα. Η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, έχει παρουσία σε αυτά τα ύδατα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία. Και βέβαια εδώ έχουμε και τις ε, ε ναυτικές ικανότητες όλων των χωρών που συμμετέχουν περισσότερο ή λιγότερο στην ε, διένεξη αυτή. Ε, έχουμε τη, το, τους διαδρόμους προσγείωσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ε, έχουμε εδώ το, υποβρύχια, ε, μαχητικά σκάφη, έχουμε τις Φιλιππίνες, έχουμε τις αγορές νέων υποβρύχιων από το Βιετνάμ, από τη Ρωσία. Εδώ δεν θα έλεγα για στρατιωτικό σχηματισμό ή ανταγωνισμό εξοπλισμό, αλλά για στρατιωτικές ικανότητες. Εδώ υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Ε, αυτό θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί. Αν δούμε τα ε, χαρακτηριστικά της Κινέζικης θάλασσας που είναι ζεστή τροπική θάλασσα, ρηχή, εκεί βλέπουμε μεγάλο αριθμό υποβρυχίων που δύσκολα μπορεί να ελιχθούν και να ε, υπάρξουν στα νερά αυτά. Οπότε μπορεί να υπάρξει μια σύγκρουση ή ένα ατύχημα που μπορεί να κλιμακωθεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ε, υπάρχουν πολλά, είναι πολλά τα διακυβεύματα εδώ. Η νότια κινέζικη θάλασσα είναι πολύ κεντρικής σημασίας. Πρέπει να πάρει κανείς θέση για την Νότια Κινέζικη θάλασσα, αν θέλει να είναι κάποιο στην περιοχή. Η αποδυνάμωση της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ε, ενέχει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Ε, συζητείται ακόμα ένας ε, κώδικας διοντολογίας ε, από το 2003 υπάρχει αλλά δεν είναι δεσμευτικός και συνεχώς υπάρχουν αλλαγές και παραδιάσεις και τέλος υπάρχει έλλειψη διακυβέρνησης, έλλειψη συνεργασίας ε, ό,τι αφορά τα καθημερινά λειτουργικά θέματα ε, ε, ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι οι χώρες αυτές χωρίς να αναδειχθεί αυτή η διένεξη ως το πρώτο εμπόδιο που βάζει τέρμα σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Βέβαια γιατί συμβαίνουν όλα αυτά θα, θα ρωτήσει κανείς. Ίσως ε, όλοι που, όσοι παρακολουθούν τη διένεξη αυτή από κοντά ή από πιο μακριά, ε, διάβασαν ένα άρθρο, ε, σε μια, όταν διαβάζουν ένα άρθρο σε εφημερίδες, το πρώτο που διαβάζει είναι τα αποθέματα υδρογονανθράκων εκεί. Αυτό είναι υπεραπλουστευμένο και παραπλανητικό ως επιχείρημα. Απλώς διότι τα αποθέματα είναι στην νότια Κινέζικη θάλασσα, αλλά ως επιτοπλίστων όχι στη διαφιλονικούμενη περιοχή. Ε, αναφέρθηκε αν οι γραμμές επικοινωνιών στρατηγική σημασία. ε, αυτές ξεπερνούν βέβαια την νότια Κινέζικη θάλασσα, ε, 5-3 εκατομμύρια ε, συναλλαγές, ε, δρόμοι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Βέβαια αυτά δεν θα πρέπει να τα ε, μπερδεύομαι. Ελευθερία στη θάλασσα και στην αυσιπλοεία υπάρχουν διαφορές. Ε, σίγουρα όμως μια, ένα ατύχημα ή μια συμπλοκή μπορεί να επηρεάσει όλα αυτά. Παρόλο που σκόπιμα εκείνα δεν θα ήθελε να διαταράξει το εμπόριο το δικό της. Επίσης, κάτι που δεν ε, είναι πολύ σημαντικό και δεν συζητείται πολύ, αλλά το ανέφερα ο κύριος Όξμαν, ε, είναι ε, η αλληλεία. Πολύ σημαντική. Το 12% των αλλιευμάτων παγκοσμίω γίνονται στην Νότια Κινέζικη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ για μια μικρή συγκριτικά περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ψαριών, 34%, ίσως και οι μεγαλύτεροι. Οι παράκτιες οικονομίες εξαρτώνται όλες από την αλληλεία, από την πρωτεΐνη των ψαριών για την καθημερινή τους διατροφή και τα αποθέματα στην νότια Κινέζικη θάλασσα σχεδόν έχουν εξαντληθεί. Σύμφωνα με κάποιες εκθέσεις, ε, το κόκκινο έχουν εξαντληθεί, τα κίτρινα όχι ακόμα και υπάρχουν και ορισμένε πράσινες είναι τα εναπομείνοντα αποθέματα ηχθείων ε, με τις κατάλληλες ελιευτικές τεχνικές, γιατί μιλάμε για εργοστάσια εδώ που λειτουργούν και επεξεργάζονται τα ψάρια, η ζήτηση αυξάνεται, ενώ τα αποθέματα ε, εξαντλούνται όλο και περισσότερο. Οπότε εδώ μιλάμε για μια μεγάλη μακροχρόνια ε, οικονομική επίπτωση που μπορεί να κρύβεται, μπορεί να αποτελεί και ε, το βασικότερο λόγο για τις εντάσεις αυτές. Πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Αυτή είναι η αντίδραση του Φιλιππινέζου Προέδρου στην ε, δήλωση της Κίνας σχετικά με την, ε, τις κατασκευές στο Σκάρμπορο βλέπετε είναι αριστερά, είναι αρκετά μεγάλη η 15 15-16 χιλιόμετρα σε μήκος, μπορούν δηλαδή να δημιουργηθούν εκεί πολύ σημαντικοί διάδρομοι προσγείωσης. Ο Φιλιππινέζος πρόεδρος είπε τι θα κάνουμε για όλα αυτά. Οι Φιλιππίνες δεν μπορούν μόνες τους να κινηθούν. Ε, ενδεχομένω ούτε μόνο είπα Μπορούμε όμως να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ενιαίο διεθνές μέτωπο που στηρίζεται στο κράτος δικαίου αλλά και στις δικαστικές αποφάσεις από το 2016. Ε, ήταν κρίμα γιατί δεν αδράξαμε την ευκαιρία ως διεθνής κοινότητα, αλλά δεν, είναι, χάθηκαν και όλα. Οι χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους ε, και να έχουν αποτελεσματική ναυτική ε, παρουσία στην περιοχή, ε, υπενθυμίζοντας τα αρχές της ναυσιπλοείας. Οι περιβαλλοντικές λύσεις είναι ένας καλός τρόπος για να προσπαθήσουμε να λύσουμε τη διαφορά ή τουλάχιστον να βρεθεί κάποια ε, βιώσιμη διακυβέρνηση και να έχουμε βέβαια και μια μεγαλύτερη προσέγγιση στα οικοσυστήματα. Η Κίνα χρησιμοποιεί την περιοχή αυτή ε, όχι μόνο για σκοπούς ε, περιβαλλοντικούς αλλά για να εδρεωθεί στην περιοχή. Έχουμε διάλογο και με την ΑΣΕΑΝ και με το Βιετνάμ για την ε, θαλάσσια συνεργασία, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην, στα καθημερινά θέματα, τα λειτουργικά θέματα ε, ασφάλειας, ε, σίγουρα στα θέματα αλληλείας που έχουμε μεγάλη ε, τεχνογνωσία ε, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε σε επίπεδο ΟΗΕ για κάποιον μηχανισμό επιβολής. Μιλάμε για τις ε, ειρηνευτικές ε, ε, επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη τεχνογνωσία μας από την προληπτική διπλωματία. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Φρανς Πολ θα το αναπτύξει αυτό περισσότερο. Σίγουρα το βασικό ζήτημα είναι οι δράσεις της Κίνας που ε, εκτιλήσονται στην ε, Νότια Κινέζικη αν δούμε, στην Νότια Κινέζικη, αν δούμε και τον Ινδικό ωκεανό, βλέπουμε ότι δεν περιορίζεται στην Νότια Κινέζικη θάλασσα. Οπότε ένα ερώτημα είναι πόσο μακριά είναι το υπερβολικά μακριά από την πλευρά της κίνησης της ε, Κίνας. σε ποιο βαθμό θα κινηθούμε με τρόπο τέτοιο ώστε να ε, διαφυλάξουμε ε, ένα διεθνές σύστημα λειτουργίας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Δ. Φραντς Πολ Φαντερ από τις κάτω χώρες. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω στην ακρόαση αυτή. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις επιπτώσεις στην ε, ευρωπαϊκή ασφάλεια των εντάσεων στην Ανατολική και Νότια Συνική θάλασσα. Τα ακούσαμε και από τον καθηγητή Όξμαν. Τι διακυδεύεται όσον αφορά την ε, διεθνή νομιτάξη, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κατάσταση για την Ευρώπη και για την ε, ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό που θα κάνω λοιπόν ε, είναι ότι θα μιλήσω για τις εντάσεις υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής και θα δούμε τι σημασία έχουν όλα αυτά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα, αν δείτε την οθόνη σας, θα δείτε διάφορες φωτογραφίες. Τις έβαλα αυτές τις φωτογραφίες για να σας θυμίσω ε, το θερμό επεισόδιο της 1ης Απριλίου του 2001 το είπε και η Εύα Πέσοβα, υπάρχει κίνδυνος πράγματι ατυχήματος. Και ένα τέτοιο σοβαρό ατύχημα έλαβε χώρα ακριβώς το 2001 και ήταν αμέσως αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του George W. Bush. Τότε ένα αμερικανικό ε, κατασκοπευτικό αεροπλάνο πήγε πολύ κοντά στην Ίσο Χαϊνάν, την Κινέζικη, και συγκρούστηκε με ένα μαχητικό Κινέζικο, το οποίο προσπαθούσε να αναχαιτήσει το Αμερικανικό αεροπλάνο, να το εμποδίσει να πάρει τις πληροφορίες που ήθελε. Κάτι δεν πήγε καλά λοιπόν και υπήρξε σύγκρουση. Έπεσε το κινέζικο, σκοτώθηκε ο πιλότος και το αμερικανικό αεροπλάνο χρειάστηκε να κάνει κάτι πολύ δύσκολους ε, ελιγμούς και να προσγειωθεί κατεπηγόντως. Υπήρξε κρίση, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών για ένα διάστημα που επιλήθηκε μετά. Ξεχάστηκε το συμβάν αυτό, γιατί μέσα στην χρονιά εκείνη είχαμε και τα γεγονότα της 11 ε, η Σεπτεμβρίου, οπότε η γεωπολιτική προσοχή απομακρύνθηκε από την Ασία και πήγε στη Μέση Ανατολή μέχρι το 2009. Τώρα αρχίζουμε πάλι και δίνουμε σημασία στα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική και Νότια Συνική Θάλασσα. Πάντως το θερμό αυτό επεισόδιο δείχνει ότι οι ατυχήματα μπορεί να συμβούν. Και η πιθανότητα να συμβεί και πάλι κάτι τέτοιο δεν είναι αυξανόμενη. Μετά το 2001 οι εντάσεις έχουν ενισχυθεί στην περιοχή, κυρίως ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας δούμε τώρα την γεωπολιτική δυναμική που επικρατεί στην Ανατολική Ασία. Το βασικό ζήτημα, το θεμελιώδες, που επηρεάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά των χωρών στην περιοχή έχει να κάνει με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως εξισορροπητική δύναμη εκτός περιφέρειας. Γιατί πρόκειται για μια ασιατική χώρα η οποία επηρεάζει τις σχέσεις και το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ της Κίνας και των άλλων κρατών της περιοχής επειδή η Κίνα αναδύεται τώρα σαν μια περισσότερο ισχυρή δύναμη από ότι οι υπόλοιπε ασιατικέ χώρες, ακόμα και από την Ιαπωνία. Η Κίνα λοιπόν αποκαλεί μια πρόκληση για την τάξη στην περιοχή, κάτι το οποίο απασχολεί και τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή, αλλά και τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες προσπαθούν να αποτελέσουν το αντίβαρο, χρησιμοποιώντας τη δικιά τους επιρροή κυρίως τον ρόλο τους σαν μεγάλο παράγοντα ασφαλείας στην περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο από πολλές ασιατικές χώρες πλην της Κίνας, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες τα καταφέρνουν στο ρόλο αυτό χωρίς να δημιουργούν καταστάσεις κρίσης ή άλλες διανέξεις. Η Κίνα ανησυχεί πολύ για την κατάσταση αυτή από πλευράς βέβαια ασφάλειας της Κίνας είναι ιδιαίτερα απειλητικό. Οι σχέσεις της χώρας αυτής με τις γείτονες χώρες να επηρεάζεται από μία δύναμη εκτός περιοχής που θεωρεί μάλιστα η Κίνα ως γεωπολιτικό αντίπαλο. Αυτή είναι η δυναμική λοιπόν στην περιοχή σήμερα. Αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση στην Ανατολική Συνική θάλασσα, όπου η Κίνα επίσης προσπαθεί να κυριαρχήσει στρατιωτικά, κάτι το οποίο βέβαια αντιβαίνει στα συμφέροντα της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Ταϊουάν, που βασίζονται στις Ηνωμένε Πολιτείες για να διορθώσουν αυτή την ανισορροπία. Ανισορροπία που από την άλλη μεριά η Κίνα την κατάσταση αυτή, το ότι δηλαδή ζητούν οι γειτονέ τη στη βοήθεια των ΗΠΑ, είναι κάτι που το βρίσκει ιδιαίτερα απειλητικό. Και την ίδια δυναμική την βρίσκουμε και στην νότια συνική θάλασσα, όπου εκεί υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν συμφέροντα ασφάλειας. Δεν πρόκειται μόνο για τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται σε εδαφικές ή θαλάσσιες διενέξεις με την Κίνα, αλλά και άλλες χώρες στην περιοχή, όπως είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα ή τα Ιουάν, γιατί πρόκειται για διόδους επικοινωνίας που έχουν στην θάλασσα αυτή, αλλά είναι και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται, όπως είναι οι Φιλιππίνες, το Μπρουνέτε, Βιετνάμ, η τα γιατι προκειται για διοδους επικοινωνιας που εχουν στην θαλασσα αυτη αλλα ειναι και Σιγκαπούρη, που τους επηρεάζει οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ασία. Τι διακυδεύεται λοιπόν τελικά στο συνδυασμό αυτό Ανατολική και Νότια Συνική θάλασσα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μια γενής αξία των θαλασσίων αυτών περιοχών και το είπε και ο καθηγητής ε, οξω νωρίτερα ότι υπάρχουν υδρογονάθρακες και σωστά είπατε κι εσείς ότι ίσως να μην πρόκειται τόσο πολύ για τους σπόρους αυτούς δρογοναθράκων, αλλά για τους ελευτικούς σπόρους που έχουν μεγάλη σημασία. Το άλλο που διακυδεύεται εκεί είναι βέβαια το δυναμικό των θαλασσιών αυτών περιεχών όσον αφορά ε, πληροφορίες και μια τεράστια γεωστρατηγική σημασία της ε, Ανατολική και Νότια Ινικής Θάλασσα. Η πρόκληση λοιπόν για τις ΗΠΑ Πολιτείες είναι μεγάλη προκειμένου να αποδείξουν ότι μπορούν να παίξουν το ρόλο τους, δηλαδή εξισορροπητική δύναμη εκτός της περιοχής. Με την κυβέρνηση Ομπάμα ήταν που αποφασίστηκε να μπει το θέμα αυτό στην πρώτη γραμμή. Να αναφέρεται ρητά και να περάσει το μήνυμα στις χώρες της περιοχής ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πρώτα απ' όλα θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν το ρόλο τους αυτό, εξωσορροπητικής δύναμης εκτός περιφέρειας για το μέλλον και προσπαθούν να το αποδείξουν αυτό παίζοντας ενεργό ρόλο στην περιοχή, στην θάλασσα αυτή, για να συνεχίσουν να επηρεάζουν το συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσα στην Κίνα και τις γείτονες χώρες. Οπότε η πρόκληση για τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι ότι πρέπει να αποδεικνύουν ότι μπορούν να φέρουν σε πέρα στο ρόλο τους αυτών. Για την Κίνα όλα αυτά αποτελούν μια ευκαιρία. Γιατί αν η Κίνα μπορεί να συνεχίσει τη σημερινή της πολιτική ε, βαθμιάς επέκτασης της ισχύω της στην θάλασσα αυτή αποδυναμώνονται οι υπόλοιπε χώρες, ενισχύει η για τον μελλοντικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, για το κατά πόσο δηλαδή θα μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν τον εξωσορροπητικό αυτό ρόλο και αν η Κίνα μπορεί να συνεχίσει να πιέζει όπως κάνει τώρα τις Ηνωμένε Πολιτείες στην ασιατική τους πολιτική, τότε αυτό τελικά θα υπονομεύσει και τον στρατηγικό ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή. Αν όμως η Κίνα δεν το πετύχει αυτό, τότε θα έχει φανεί από τις Ηνωμένε Πολιτείε ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες να εξακολουθούν να διασφαλίζουν προστασία των χωρών της περιοχής και θα ενισχύσει αυτό και τις διμερείς του σχέσεις με τι άλλες χώρες στην Ασία. Για την Ιαπωνία, ο ρόλος της, ο γεωστρατηγικός, είναι μεγάλη σημασία για το μέλλον. Γενικότερα στην περιοχή και όχι μόνο εξαιτίας της Κίνας, μένει λοιπόν να δούμε τι θα κάνει η Ιαπωνία στο μέλλον. Δεν είναι σαφές ακόμα τι θα έκανε η Ιαπωνία αν εγκατέλειπε την σημερινή τη σημαντική αμυντική εξάρτηση βάσει της συμφωνίας που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ αναφέρω πέντε σενάρια, πέντε δυνατότητες. Η μία θα ήταν η Κίνα να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις της ή να τις περιορίσει. Αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται να υλοποιείται, γιατί να δεν δείχνει σημάδια ότι θα εγκαταλείψει ή θα περιορίσει τις διεκδικήσεις της. Το δεύτερο σενάριο θα ήταν να αποσυρθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, να αποφασίσουν να αποσυρθούν από την περιοχή. Προς το παρόν και αυτό φαίνεται να πραγματοποιείται γιατί για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντική περιοχή, γιατί δεν έχει να κάνει τελικά μόνο με την Ανατολική Ασία, οπότε δεν είναι ένα λιθοφανές σενάριο. Έπειτα η στάση του Πρόεδρου Τραμπ δεν δείχνει να οδηγηθεί σε κάτι τέτοιο. Προς το παρόν δείχνει ότι επενδύει πολύ στην Αμερικανική στρατιωτική δύναμη. Συνεπώς θέλει να χρησιμοποιήσει την δύναμη αυτή περισσότερο και έπειτα παίρνει πολύ στα σοβαρά τις οικονομικές σχέσεις της Αμερικής με την Κίνα. Συνεπώς και γεωπολιτικά και στρατιωτικά για τις Ηνωμένε Πολιτείε το σενάριο είναι ότι μάλλον θα ενισχύσει τις ε, σχέσεις με την περιοχή παρά το αντίθετο. Το τρίτο σενάριο θα ήταν η κοινότητα του ειρηνικού. Αυτό είναι κάτι που το είχε χρησιμοποιήσει ο Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίο είχε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινότητα του ειρηνικού με την Κίνα, τι Ηνωμένε Πολιτείε και του άλλου παράγοντε στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτό το τρίτο είναι που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά και πάλι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό το σενάριο θα πραγματοποιηθεί. Το τέταρτο θα ήταν να συνεχιστεί απαόριστο το status quo. Είναι και το πιο πιθανό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι σαφές το κατά πόσο όντω επαόριστο θα μπορεί να συνεχιστεί, γιατί ο συσχετισμός δυνάμεων καθημερινά αλλάζει. Η Κίνα αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη όσο περνά ο καιρό Και παρά τι προσπάθειες που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ιδίως από το 2009 και μετά, η αβεβαιότητα που επικρατεί μεταξύ των ασιατικών χωρών για το μέλλον της γεωπολιτικής τάξης είναι κάτι που συνεχίζεται και αυξάνεται. Και το τελευταίο σενάριο θα ήταν μια σύγκρουση ή ένας μεγάλος πόλεμος ή μια περιορισμένη σύγκρουση. Δεν φαίνεται να συμβεί αυτό σύντομα, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Συνεπώς, μια περίοδος αυξανόμενων εντάσεων είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να καταλήξει σε κάποιο είδου σύγκρουση. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι εντάσει στην περιοχή ήδη επηρεάζουν την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ασφάλεια. Λάβουμε υπόψη μας επίσης την οικονομική ε, δύναμη της Κίνας που δεν είναι ενισχυόμενη ανά τον κόσμο. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την πρωτοβουλία της Κίνας One Belt, One Road, ενιαία ζώνη, ενιαία διέλευση, που σημαίνει ότι θέλει η Κίνα να επεκτείνει την επιρροή της και τη διπλωματική δυτικά, βοηθώντας την Ευρασία και μέρος της Αφρικής να δημιουργήσουν μεταξύ τους μια ολοκληρωμένη οικονομική ζώνη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κίνα ενισχύει την οικονομική της επιρροή στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο περνά ο καιρός σε σχέση με την γεωπολιτική της θέση εξομοιούται με τις χώρες ΑΣΑΝ, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι πολύ ευνοϊκό για την Ευρώπη. Και αν δούμε την επιρροή που μπορεί να έχει η Κίνα είναι σημαντικό να προσέξουμε το δυναμικό, πώς ε, δημιουργούνται οι σχέσεις μέσα στην ΑΣΕΑΝ. Η Κίνα θέλει να έχει οικονομικές σχέσεις με κάποιες χώρες μεταξύ των ΑΣΕΑΝ, ώστε όταν θέλει να δράσει σε θέματα ασφάλειας στην περιοχή να μπορεί να τις έχει με το μέρος της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο. Έχουμε 28 χώρες μέλη. Κάποιες έχουν ισχυρές οικονομίες, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλλά υπάρχουν άλλες που δεν είναι τόσο δυνατές οικονομικά. και έχουν ή θα αναπτύξουν πολύ στενές σχέσεις με την Κίνα. Η διαδικασία αυτή θα καταστήσει πιο δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ενιαία. και τελικά μπορεί, αν όχι να παραλύσει, αλλά τουλάχιστον να καταστήσει πολύ πιο δύσκολη τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Ανατολική και Νότια Συνική Θάλασσα. Κάτι το οποίο θα δημιουργήσει εντάσεις, δυσπιστία μεταξύ πρώτα των ευρωπαϊκών χωρών μελών και δεύτερον μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, κάποιες άλλες επιπτώσεις για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν υπάρξει κάποια σύγκρουση είτε μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας είτε μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι άμεσες επιπτώσεις φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις προβλέψει κανείς. Αν υπάρξει μια μεγάλη σύγκρουση φυσικά θα υπάρξουν τεράστιες σε συνέπειες. Έμεσα όμως, ακόμα και αν η σύγκρουση δεν είναι μεγάλη, αλλά τοπική, με την εμπλοκή και των ΗΠΑ και της Κίνας, οι επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι μεγάλες. Ένα τέτοιο σενάριο με τέτοια ιδέα αναπτύχθηκε σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και μπήκε σε ιστοσελίδα μάλιστα που ανακοίνωνε και την ακρόαση αυτή. Τι θα μπορούσε να γίνει τότε. Επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε σε μια τέτοια περίπτωση κρίσης θα ήθελε να διευθετήσει την κρίση αυτή, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν νέο συσχετισμό και συμπεριφορά σε άλλες περιοχές όπως είναι η Ανατολική Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και αυτό θα επηρέαζε κυρίως αν αυτές οι άλλες περιοχές αντιλαμβανόντουσαν ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είτε μπορούν να αντιμετωπίσουν την Κίνα και να προστατεύσουν τους εταίρους τους ή από την άλλη μεριά να αποδειχτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ανάλογα αυτό θα δημιουργούσε οπορτουνιστικές ή όχι τάσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχουμε δύο εισηγητές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων παρόντες. Ο κ. Κόφερ πρώτα απ' όλα που είναι ο μόνιμος εισηγητής για την Νοτιοανατολική Ασία και μετά ο κύριος Μπέλντερ, εισηγητής για την Κίνα. Προτείνω λοιπόν Κύριοι, να πάρετε το λόγο και αν μπορείτε παρακαλώ να περιοριστείτε σε δύο λεπτά ο καθένας. Ας ξεκινήσω, να μου επιτρέπετε κύριε Μπέλτερ. Ο κύριος Μπούτι Χόφερ είναι ο μόνιμος ε, εισηγητής. Άρα προηγείται ο κύριος Μπούτι Χόφερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να επενθυμίσω σε όλους ότι αυτό το κοινοβούλιο κατά το παρελθόν ήδη ψήφισε ένα κείμενο καλώντας όλα τα μέρη στην ε, διαφορά αυτή στην Νότια Συνική Θάλασσα να σεβαστούν την απόφαση του πάνελ του Άγκρος. Το ψηφίσαμε αυτό πριν ληφθεί η απόφαση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο διατύπωσε σαφώς την άποψή του για το ζήτημα. Δεύτερον, Είμαι ευγνώμων προς τους εμπειρογνώμονες για τις ε, παρουσιάσεις τους. Πρέπει όμως να πω ότι θλίβομαι κάπως, διότι βλέπω διάκριση, διαφορά μεταξύ αυτού που περιγράφεται σε σχέση με τα όσα έκαναν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως το Συμβούλιο, διαμορφώντα την πολιτική τους. Δεν ήταν εκεί η καλύτερη στιγμή της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Χρειαστήκαμε περίπου δύο μέρες. Και θα συμφωνεί και ο Σβίγκαν με αυτό. Μας πήρε δύο μέρες, λέγω, για να προβούμε σε μια δήλωση που λέει ότι παραδεχόμαστε την ισχύ, αναγνωρίζουμε την απόφαση. Ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα όταν σε μια διπουργική σύνοδο ΑΖΕΑΝ Ευρωπαϊκής Ενώσεως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με μια διατύπωση του ΑΖΕΑΝ που συμπεριλάμβανε την Καμπότζη και το Λάος ε, που είναι ουσιαστικά πελατειακά κάτι ενάντια της Κίνας και είχαν προτείνει αυτές οι χώρες ε, ε, μια διατύπωση Αυτή είναι μια σύγκρουση πολύ σημαντική θα έλεγα με μεγάλες συνέπειες και σε πρόσφατες συνομιλίες που έχω σε διάφορες πρωτεύουσες περιοχές πρέπει να σας πω ότι είδα ότι η στάση που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι καταδικάστηκε ε, σε περισσότερες περιπτώσεις. Οι συνομιλητές μου μου είπαν ότι αισθάνθηκαν ότι ε, αφέθηκαν, ότι παραμερίστηκαν, ότι αγνοήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Χαίρομαι που οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την βραχονισίδα Σκάρμπορο αναφέρθηκαν. Είναι άλλη, άλλο ένα όριο αυτό, μια κόκκινη γραμμή, που χάραξε κάποιος στην αμμουδιά και τη λησμόνησε. Και οι Κινέζοι αποφάσισαν να περάσουν αυτή τη γραμμή. Τώρα να εκνευριζόμαστε μέσω ρητορική δεν έχει νόημα αν δεν συμφωνούμε μεταξύ κρατών μελών. Δηλαδή να πούμε ότι είμαστε τουλάχιστον μια ένωση που υποστηρίζει το διεθνές ε, δίκαιο, τη διεθνή ένωμη τάξη και πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας αυτή σε συγκεκριμένε ε, αντιδικίες όπως αυτή και σε συγκρούσεις. Είναι πολύ επικοδομητικό το ότι τίθεται το ζήτημα στην Υπεπιτροπή μας αυτή. Ελπίζω να βρούμε κάποιους τρόπους να πείσουμε τους συναδέλφους μας, τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτως ώστε να ασκήσουν πιέσεις επί κυβερνήσεων των κρατών μελών. Διότι οι κυβερνήσεις τελικά υπολείπονται των ενδεωδών και των ελπίδων των εταίρων μας ε, στην Νοτιοανατολική Ασία. Ευχαριστώ, κύριε. Ο κύριος Μπέλντερ, που είναι ο εισηγητής ε, που είναι αρμόδιος για την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Χαίρομαι για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε από τους ειδικού εδώ. Και για να αρχίσω θέλω να υπορρομήσω αυτό που είπε και ο συνάδελφος Μπάτι Κόφε. Η κυρία Πέσοβα αναφέρθηκε για την παρουσία των Γάλλων στην νότια Συνική θάλασσα. Και άλλες χώρες ε, μέλη του ζητήθηκε ε, συμβολικά έστω να προσφέρουν ε, κάποια δύναμη εκεί. Και η Κίνα είπε όχι. Ρωτάω λοιπόν τι έχει γίνει τελικά με αυτά. Ξέρουμε. Πέρσι υπήρξε και μία μελέτη ε, σχετικά με το πόσο ενωμένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το συμπέρασμα ότι δεν είναι, είναι κατακαιρματισμένη. Οπότε θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα ποιες είναι οι αντιδράσεις των χωρών μελών μετά την έκκληση που έγινε το 2016 από τη Γαλλία προκειμένου να παρευρεθούν δυνάμεις και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην περιοχή που εξετάζουμε. Έχω και την μελέτη αυτή ενός πολιτικού ιδρύματος για την περιοχή περί τίνος πρόκειται, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και στο τέλος της μελέτης αυτής λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την τήρηση του δίκαιου της θάλασσας, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και ρωτάω πώς μπορούμε να αποφύγουμε την κλιμάκωση και πώς μεσοπρόθεσμα θα μπορούσε να, ε, να ζητήσει να υπάρξει μία διάσκεψη για την περιοχή αυτή, παίρνοντας βέβαια κάποιες αποστάσεις από τους ε, κύριους παίκτες, την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείες και βέβαια προστατεύοντας τα δικά μας τα συμφέροντα, αποκλιμακώνοντας την ένταση, αντί να αφήσουμε την υπόθεση μόνο στην Κίνα και στις άλλες χώρες της περιοχής. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Πάντως ε, προβληματίστηκα από αυτά που είπατε, που άκουσα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, colleague. And, uh, Ευχαριστώ συνάδελφε. Και άλλοι δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Τσάρλς Τάνοκ πρώτα απ' όλα. Uh, thank you, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ καλά αυτά που είπατε κύριε Μπουτεκόφερ. Φοβούμαι όμως ότι παρόλο που πιστεύω στην πολύπλευρη και πολυσχεδή προσέγγιση και πρέπει να επικρατεί και το κράτος δικαίου σε διεθνές επίπεδο είναι σαφέστατο όμως ότι η Κίνα αγνόησε πλήρως την απόφαση του δικαστηρίου του Άγκλος όσον αφορά το ζήτημα και θα εξακολουθεί να αμελεί και να αγνοεί το διεθνέ δίκαιο όταν της, τη βολεύει. Και το λέω με βαθιά θλίψη αυτό που λέω. Με, ε, ε, Πιστεύω ότι η Βρετανία μετά το Brexit δεν θα θέλει να ασκήσει πίεση στην Κίνα, διότι θα θέλει να συνάπτει διμερείς συμφωνίες ε, με την Κίνα. Όταν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι προβληματικές εμπορικά αν οι διαπραγματεύσεις πάνε άσχημα. Και είδαμε μια απαρχή της προσεγγίσεως με, με τον George Osborne, με την προηγούμενη κυβέρνηση. Ε, δεν βλέπω τώρα η χώρα μου, κυρίως μετά το Brexit, να είναι ιδιαίτερα πρόθυμη να αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πίεση πολυπλεύρος και να λύσει το θέμα. Το λέω αυτό με θλίψη, αλλά αναλύω τα γεγονότα. Όποτε με ρωτούν για το θέμα της ραχονισίδας Κάρμπορο, η τυπική ε, απάντηση είναι ότι θα το αντιμετωπίσει Άζαν σε κάποια σκοτεινή επιτροπή. Άλλη ερώτηση έχω. Εδώ μιλούσαμε για την ε, νοτιοτολική θάλασσα της Κίνας. Εγώ ήμουν ο πρόεδρος των φίλων της Ταϊβάν και είμαι επίτιμο πρόεδρο ακόμα. Και η Ταϊβάν ενδιαφερόταν πολύ σε αυτή τη διαφορά, τη διένεξη για τη Νότια Συνική Θάλασσα, διότι ανήκει, ε, έχει και αξιώσει για τα Σενκάκου ε, νησιά. Ήταν υποτίθεται θέμα σύνοϊαπωνικό, αλλά ενδιαφέρεται και η Ταϊβάν. Διότι ιστορικός και παραδοσιακός ήταν ταϊβανέζικα νησιά, ειδικούνται από την Ταϊβάν και όχι από την υπηρετική Κίνα και ενδιαφέροντα. Ο πρώην πρόεδρο τη Ταϊβάν, τον οποίο συνάντησα δύο φορές όταν επισκέφθη την περιοχή, έγραψε ένα σύγγραμμα και το ανέφερα εγώ σε κάποιο άρθρο. Εκεί τα Κάγκοτζα Γιουκάι ε, τα παρουσίασε, βρήκα τη λύση σύμφωνα με τη συμφωνία με την, ε, όπως έγινε για την Ανταρκτική, όπου αφέθηκαν εκτός ε, διάφορες εδαφικές διεκδικήσεις και αναπτύχθηκαν οι εκμεταλλεύσεις ε, όπως αφορά την αλληλεία και τα ορυκτά με κανονικό φυσιολογικό τρόπο. Το είχα πενέσει σαν προσέγγιση τότε και στο Κοινοβούλιο και υπό την ιδιότητά μου σαν πρόεδρος της ομάδας φιλίας για την Ταϊβάν αλλά αυτό δεν προχώρησε. Αυτή η έννοια, δηλαδή να δούμε τι γίνεται με άλλες αμφισβητούμενες περιοχές όπως η Ανταρκτική που είναι πλουσιότατες σε φυσικούς πόρους, αλλά που τη διεκδικούν πολλές χώρες, κομμάτια της περιοχής, και όμως συνεργάζονται επιστημονικά και διεξάγουν έρευνα και αφήνουν τις διεκδικήσεις εκτός. Θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση πολυμερής. Αλλιώς, σε κάποια φάση κάποιος θα πατήσει την άρκη και θα ξεσπάσουν οι ε, εχθροπραξίες. Ναι, μπορώ να υπογράψω και εγώ, να προσυπογράψω εγώ στην ερώτησή σου, Τσάλς. Ακριβώς αυτό το ερώτημα ήθελα να θέσω. Ε, κανένα πρόβλημα. Ναι, εντάξει, τι μοιραζόμαστε, μοιραζόμαστε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει το λόγο. Είπατε προηγουμένως ότι ε, οι Κινέζοι κάνουν επενδύσεις σε κάποιες αδύναμες ευρωπαϊκές οικονομίες και οι οποίες μπορεί στο μέλλον να δυσχεράνουν μια ε, συνολική ε, ευρωπαϊκή αντιμετώπιση ε, της ε, κινέζικης επέκτασης οικονομικά ή κάποιων προκλήσεων ή διενέξεων. Σε ποιες ακριβώς επενδύσεις αναφέρεστε. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι αν μπορείτε να μας πείτε δύο στοιχεία κατά πόσο γνωρίζοντα τα προβλήματα που υπάρχουν ε, στην νότια και ανατολική Κινέζικη θάλασσα, προχωράει η επένδυση ε, που αφορά την ε, χερσαία δίωδο του δρόμου του μεταξιού. Πώς πάνε αυτές οι επενδύσεις. Thank Σας ευχαριστώ. Και έχω άλλη μία ερώτηση απευθυνόμενη βασικά προς τον κύριο Βίλαντ αλλά και την απευθύνω και προς τους άλλους δύο διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους μας μαθήματα που μάθαμε. Υπάρχει κάποιο μάθημα που μπορούμε να συνάγουμε από την εμπειρία μας όσον αφορά την επιτυχέστατη αποστολή επιχείρηση Αταλάντη και τους εξωτερικούς εταίρους που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή μέσω ενός ειδικού μηχανισμού σε είδε από ό,τι θυμάμαι υπάρχει κάποια ομοιότητα που μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτό που πρότεινε και ο Μπέλντερ να το λάβουμε υπόψη ίσως κάπως αυτό μπορούμε να το παρουσιάσουμε ήταν ένας πολύ καλός τρόπος επίλυσης πολύ δύσκολων προβλημάτων. Με πλήρη σεβασμό των διαφορών που επικρατούσαν, όμως ήταν μοναδική εμπειρία. Θα ήθελα όλα τα μέλη του πάνελ εάν είχαν την καλοσύνη να απαντήσουν στις ερωτήσεις που έθεσαν οι ευρωβουλευτές μας. Με την ίδια σειρά παρακαλώ, ο κύριος Βέγκαν και μετά ο καθηγητής Χάξμαν, μετά η κυρία Πέισοφα και ο κύριος Βαντερπούτεν. Ο κύριος Βέγκαν. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να τονίσω καταρχήν ότι Αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποστηρίζει απόλυτα την απόφαση της ΟΥΝΚΛΟΣ και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όταν δεν είχε έρθει ακόμα ο κ. Μπιουτικόφερ, είχα την ευκαιρία να διαβάσω ένα κομμάτι από τη διακήρυξη των 28 από πέρσι το Μάρτιο, όπου εκφράστηκε σαφής ανησυχία και τονίστηκε η σημασία ε, και η, Σιμόρ, της απόφαση Σούγκλος και η, ε, ο σεβασμός της και η εφαρμογή της. Ε, εμείς ε, καλωσορίσαμε τη διεθνή δικαιοδοσία. Η αναγνώριση δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαφοροποίηση από την ε, δικαιοδοσία από αυτή την απόφαση και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται ε, από τις αρχές του διεθνούς δικαίου της Ούγκλος και είναι υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Μην ε, υπάρχει αμφιβολία λοιπόν σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σίγουρα δεν αναστέλει τις σωστές διαδικασίες η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού τάσεται υπέρ της Ούγκλος για τις διαδικασίες επίλυσης διεθνών διαφορών. Είπα και πριν ότι έχουμε πάνω από το 40% του ε, διεθνούς εμπορίου μας που περνά από την ε, αμφισβητούμενη αυτή περιοχή που συζητάμε. Τώρα, στην ερώτηση του κυρίου Μπέλτερ. Δεν συγκαλούμε συχνά ε, διασκέψεις ειρήνης, βέβαια για τη Συρία, το Αφγανιστάν, η Συρία θα γίνει σε λίγες μέρες μάλιστα. Εδώ όμως θέλουμε να βοηθήσουμε τα μέρη. Χαιρετίζομαι την ε, επιβεβαίωση από ΑΖΕΑΝ και Κίνα ότι γίνονται συνομιλίες για κώδικα δεοντολογίας ε, σύμφωνα με τα πρώτα του 2002. Αυτό δεν το κάνουμε λόγω των οικονομικών μας μόνο συμφερόντων στην περιοχή. Το κάνουμε γιατί δεσμευόμεθα από την Ούγκλος, όπου όλα μας τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος. Έχουμε επίσης συμφέρον από την ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ασίας αφού το 2012 ως Ευρωπαϊκή ε, ένωση ε, προσχωρήσαμε στη συμφωνία του 76 για την ειρήνη και συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ασία και αυτό ε, ενέχει νομικά δεσμευτικές δεσμεύσεις για όλα τα μέρη. Εμείς συγκεκριμένα στηρίζουμε τις συνομιλίες και αν προσκληθούμε θα κάνουμε παρουσίαση. Η ΑΖΕΑΝ και η Κίνα αυτή τη στιγμή θέλουν να κάνουν συνομιλίες μεταξύ τους μόνο. Ε, με την ΑΖΕΑΝ όμως ε, έχουμε σεμινάρια υψηλού επίπεδου για την θαλάσσια ασφάλεια. Το τελευταίο έγινε το Ιούνιο του 2016 το, στο Βιετνάμ ως μέρος μέτρων ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα μέτρα αυτά θα συνεχιστούν και μπορεί να κάνουμε κάτι παρόμοιο με την Κίνα ίσως στα πλαίσια του Περιφερειακού Φόρουμ ε, του Ασιατικού. Οι εμπειρίες που αναφέρατε κυρία Πρόεδρε έχουν σημασία η στενή συνεργασία για τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος αλλά και για να έχουμε κοινή διαχείριση των πόρων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και η Ευρώπη έχει ειδική συμβολή να δώσει που δεν είναι πρωτίστως η σημαία και οι ναυτικές τα, σκα, τα, τα σκάφη αλλά μια σωστή κοινή διαχείριση. Τα εδαφικά ζητήματα, τα θέματα χωρικών υδάτων θα πρέπει να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο για κάθε περίπτωση χωριστά. Τέλος, να πω ότι εκείνοι που επικρίνουν το αποτέλεσμα των διαδικασιών στο Συμβούλιο πρέπει σίγουρα να εξετάσουν τα εθνικά συμφέροντα του κάθε κράτους μέλους μας. Αν δούμε όμως την αντίδραση εταίρων όπως Καναδάς, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, ΗΠΑ, θα δείτε ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, είναι στο μέσον, δηλαδή έχει μια μετριοπαθή επιλογή ε, όρων. Εμείς ε, ωφεληθήκαμε από την απόφαση Ούγκλος και τις ε, αποκλειστικές οικονομικές ζώνες που είναι περίπου 20 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια περιοχή πολύ μεγαλύτερη από την, ε, το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προφανώς η τελευταία απόφαση ήταν ε, απόφαση ορόσημο γιατί καθόρισε τα χαρακτηριστικά για την ύπαρξη ε, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ευχαριστώ πολύ, Διευθυντά Βίγκαντ, και τώρα δίνω το λόγο στον καθηγητή Όξμαν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, κάποια σχόλια. Πρώτα απ' όλα, προσοχή, προσοχή στην τάση να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο θαλάσσιο εμπόριο και την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μία από τις ιστορικές λειτουργίες της ελεύθερης ναυσιπλοείας ήταν πάντα η προστασία του θαλάσσιου εμπορίου από την ε, επιρροή είτε χωρών είτε ε, ιδιωτικών ε, παραγόντων όπως για παράδειγμα την πειρατεία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί λοιπόν όταν ζητούμε αυτή τη διαφοροποίηση. Φυσικά πάντα οι χώρες έχουν τα δικά τους συμφέροντα στο θαλάσσιο εμπόριο. Έχουν όμως και την τάση να προσπαθήσουν να προστατεύσουν το δικό τους εμπόριο σε βάρος των ανταγωνιστών τους. Οπότε, πού θα φτάσουμε με μια τέτοια κατάσταση. Αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με το Γιβραλτάρ και τις διεκδικήσεις τότε των ε, Ισπανών. Το δεύτερο, και βέβαια εντάξει το ξέρω ότι η ζωή δεν είναι απλή και εύκολη, αλλά το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι για κάθε χώρα στην περίπτωση αυτή ισχύει το ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα ουσιώδη συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, και του ρόλου που θα μπορούσε να παίξει προκειμένου να συνεισφέρει σε μια φιλική διαθέτηση. Εγώ θα περιοριστώ σε αυτά. Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει και τους δύο ρόλους. Αλλά, το ξαναλέω, προσοχή γιατί αν ακολουθήσουμε αποκλειστικά την άποψη που λέει ότι θα μπορούσε να συμπεριφερθεί σαν αυτόν που προσπαθεί να συμφιλιώσει, μπορεί τελικά να έχει σαν αποτέλεσμα επί της ουσίας να μην μπορέσει να επηρεάσει τα πράγματα. Ξέρω ότι δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα και ούτε λέω ότι εγώ είμαι σε θέση να το λύσω εδώ. Αλλά κάτι ακόμα. Είναι πολύ χρήσιμο να σκεφτούμε πολλά και διάφορα μοντέλα που επιτρέπουν στις χώρες να διεκδικήσουν νομικά τις ε, αξιώσεις τους. Ακόμα και αν τηρούσε την απόφαση, τη ευόταν η Κίνα, που έχει μεγάλη επίπτωση και στα Spartles, γιατί γι' αυτά δεν τίθεται θέμα 12 μιλίων, Επιπλέον υπάρχει και μια νομική υποχρέωση για συνεργασία επειδή πρόκειται για μια μη στη θάλασσα. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τα μοντέλα. Δεν λέω ότι πρέπει να προσδεθούμε σε ένα ή άλλο μοντέλο, αλλά να τα έχουμε υπόψη μας όλα. Ελπίζω να βοήθησαμε αυτό. Πρόεδρος, θέλω να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε στη διάθεσή μας πόσο. 12 λεπτά λέει η πρόεδρος. Και μετά οι διερμηνείς θα φύγουν. Αυτό συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε ευγνώμονες στους διερμηνείς για το έργο τους, αλλά αυτό ισχύει. Λοιπόν, η κυρία Πέσοβα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Για την παρατήρηση του κυρίου Μπαϊτικόφερ συμμεριζόμαστε την απογοήτευσή σας και καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο σκληρή δουλειά έγινε πριν φτάσουμε στη δήλωση αυτή. Αλλά για κάπως πιο θετικά. Αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι έχουν υπάρξει και προηγουμένως δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την δικαστική απόφαση αλλά και από τη διάσκεψη κορυφής των G7 και τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στην Ιαπωνία, όπου συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τα θυμηθούμε και αυτά όταν μιλάμε για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα για τις κοινές εξελίξεις. Συμφωνώ με τον καθηγητή Όξμαν για την νομική υποχρέωση να συνεργάζονται οι χώρες που είναι σε στη θάλασσα και για την συνεργασία για τους ε, πόρους της περιοχής όσο περιμέναμε τη δικαστική απόφαση. Είναι αλλιώ ε, στην Αντακτική στην Ευρώπη. Υπάρχει πρωτοβουλία για την ειρήνη στη Νότια και Ανατολική Συνική Θάλασσα. όσον αφορά τέτοιες διενέξεις για την Ανατολική Συνική Θάλασσα υπάρχουν ε, περιοχές που αναπτύσσονται από κοινού ε, joint seismic undertakings κάποιοι είδους κοινοπραξίες και όσοι συμμετέχουν το έχουν εξετάσει αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Υπήρξαν πρωτοβουλίες για εργαστήρια στην Ινδονησία αλλά και στον Καναδά προκειμένου να πετύχουν τον χαμηλότερο δυνατό κοινό παρονομαστή. Το θέμα με τις joint developments είναι πώς αρχίζει η συνεργασία. Αν ορίσουμε τις χώρες, πού θα γίνει η συνεργασία. Στην περίπτωση της νότιας συνικής θάλασσας, το ένα ήταν ότι κάποιοι λέγανε όχι αυτό δεν είναι διαφιλονικούμενο, είναι δικό μου. Και τελικά είναι χάσιμο χρόνου, πόρων, ενέργειας. για τη συμβολική παρουσία. Ευχαριστώ κύριε Μπέλντερ για την ερώτησή σας. Όπως γνωρίζετε, πέρυσι και οι Υπουργοί Άμυνας αναφέρθηκαν στη δυνατότητα αυτή. Η ιδέα παραμένει στο τραπέζι, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το που βρίσκεται η Γαλλία σήμερα. Η Ιαπωνία θα επισκεφθεί την Γαλλία και ίσως να συζητηθεί αυτό. Και δεν πρέπει να το αφήσουμε στην πάντα Σίγουρα είναι λεπτό. Θα ήμουν η πρώτη που θα υποστήριζα μια τέτοια πρωτοβουλία για την Αταλάντα. Έχετε δίκιο κυρία Πρόεδρε. Ήταν επιτυχής επιχείρηση η Αταλάντα. Είναι μια αποστολή και έπα στη θάλασσα. Και η διεθνής κοινότητα παρατηρεί πολύ προσεκτικά τι γίνεται. Και όταν μιλάμε για την εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αταλάντα, μιλάμε πρώτα απ' όλα. Το θέμα της πειρατείας είναι κάτι ουδέτερο, γιατί δεν πρόκειται για κάποια χώρα. Το νομικό πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό. Αν μπορούμε να έχουμε μια αποστολή ΚΕΠΑ για την ελευθερία ναυσιπλοείας, βεβαίως θα ήταν ιδανικό. Πρόεδρος, για να διευκρινίσω, εγώ δεν σκεφτόμουν αποστολή ΚΕΠΑ, σκεφτόμουν έναν ειδικό μηχανισμό που θα συνοδεύει την Αταλάντα για να επιτευχθεί η συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους διευκολύνοντας, βοηθώντας την ελευθερία αναψυπλοίας για εμπορικούς λόγους. Για εμπορικούς λόγους. Αυτό μας είπε και ο κύριος Σόξμαν. Έτσι, στο περιθώριο. Ναι, ναι, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να εξετάζουμε. Ο κύριος Βαντερπούτεν τώρα. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο από τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, το ερώτημα του κυρίου Μπέλντερ, που αφορά τον ευρωπαϊκό ρόλο για τη διοργάνωση μιας κάποιας ειρηνευτικής διάσκεψης. Η ιδέα να μαζευτούν τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συζητήσουν τα ζητήματα που δημιουργούν εντάσεις και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια σύγκρουση στο μέλλον, αυτή καθεαυτή θα μπορούσε να έχει μεγάλη συμβολική αξία, κυρίως συμβολική. Δεν θα είναι εύκολο, πιστεύω, να πιστούν τα μέρη να συμβάλλουν ή να συμμετάσχουν. Ξεκινώντας από την Κίνα. Είναι πολύ ευαίσθητη για εξωτερική παρέμβαση, για μη περιφερειακούς παίκτες και για μη διμερείς επίσης ε, βάση συζητήσεων. Όμως ε, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσπαθήσει να προτείνει κάτι τέτοιο. Όμως είναι σημαντικό πιστεύω να σκεφτούμε το ευρύτερο πλαίσιο της προσεγγίσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο βασικός στόχος, η βασική προσανατολισμή που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θέλει να προωθήσει κάποια πρωτοβουλία. Δύο σαφείς προσανατολισμοί είναι οι εξή. Πρώτα απ' όλα να διατηρηθεί το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θα έλεγα να προσπαθήσει να τονώσει, να ενθαρρύνει τα μέρη να κινηθούν προς το τρίτο ενδεχόμενο του καταλόγου μου, το τρίτο σενάριο. Δηλαδή μια κοινότητα του ειρηνικού όπου εκεί η θα αλλάξουν το ρόλο τους σαν εξωτερικός φορέας, αποστατιωτικό, μάλλον σαν εξωτερικός φορέας, να παίζει ρόλο διπλωματικό και όχι στατιωτικό. Και Κίνα να αλλάξει συμπεριφορά και να αποκλιμακώσει τις αξιώσεις της, που είναι επιβλαβής ε, για τα συμφέροντα των μικροτέρων γειτόνων της. Προφανώς, όπως προανέφερα, είναι πάρα πολύ δύσκολος στόχος. Όμως να καθοριστεί αυτός ο μακροπρόθεσμος στόχος θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε ε, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω σχετίζεται με τι άμεσε επενδύσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη, κινέζικες επενδύσεις που σχετίζονται με τη μία ζώνη, μία διαδρομή ή το νέο δρόμο του, ε, του μεταξιού. υπάρχουν περιφερειακές διαφορές. Κυρίως όσον αφορά το νέο δρόμο του μεταξύ, Εστιάζεται στην νοτιοανατολική Ευρώπη, Ελλάδα και Βαλκάνια. Εκεί συγκεντρώνεται η Κίνα. Αλλά και στις κέντροευρωπαϊκές χώρες, ανατολικές χώρες Ευρώπης και νότιες χώρες Ευρώπης. Τούτου λεχθέντος, είναι ακόμα πιο σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στο τέλος πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσουν πολύ στενές και σημαντικές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα. Αυτό που λέω δεν αφορά τόσο πολύ τις ξεχωρικές περιπτώσεις άμεσων επενδύσεων, αλλά την όλη ιδέα, σύμφωνα με την οποία ότι λόγω του αυξανόμενου ρόλου της Κίνας ως επενδυτού και οικονομικού εταίρου, όλα τα, έναντι όλων των ευρωπαϊκών καταμελών, τελικά θα είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην λαμβάνει υπόψη αυτές τις οικονομικές εξαρτήσεις. Και θεωρώ ότι διάφορες χώρες έχουν και διαφορετικά οικονομικά ζητήματα και συμφέροντα που διακυβεύονται σε διάφορες χρονικές στιγμές. Άρα είναι πολύ δύσκολο και 28 χώρες να βρουν κοινή θέση λόγω αυτών των εσωτερικών διαφοροποίησεων. Ευχαριστώ κύριε Βάντεμπούτεν. Κυρίες και κύριοι, φοβούμε ότι ο χρόνος μας έληξε, πάει η χρονοθυρίδα μας, οπότε ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ για την συμμετοχή τους σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι είναι απλώς η απαρχή των συζητήσεών μας όσον αφορά την Νοτιοανατολική Ασία και όλος ιδιαίτερος όσον αφορά τις εντάσεις στην νοτιοανατολική ε, Κινέζικη θάλασσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση, καθώς και τους διερμηνείς. Εμείς ευχαριστούμε την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ. Να είστε παρόντες αύριο. Και επίσης έχουμε αύριο μια συνεδρίαση της ΣΕΝΤΕ, μόνο το πρωί, μέχρι τις 12.30. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.